Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε την επανέναρξη της ε, συζήτησης. Υπάρχουν ε, τα πρακτικά της χθεσινής ε, συνεδρίασης. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, άρα εγκρίνονται τα πρακτικά. Πρώτο σημείο στη μερίσια διάταξη.